Σάνμπερκ για ε, το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Επειδή φεύγω τον Ιούλιο από αυτό το Κοινοβούλιο, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχω απόψεις για το πρόγραμμα του Κοινοβουλίου για το 2010 αλλά θα πρόδιδα αυτούς οι οποίοι με έστειλαν εδώ τα τελευταία δέκα χρόνια αν δεν χρησιμοποιούσα τη δυνατότητα που μου δίνεται να διαμαρτυρηθώ για τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Είναι σκανδαλώδης ε, δαπάνη και κατάχρηση των χρημάτων των φορολογουμένων. Υπάρχουν κτίρια στις Βρυξέλλες και όταν συναντώ πολίτες από το Ηνωμένο Βασίλειο τα έξοδα και ο κόπος που ξοδεύονται γενικά που προκαλούνται από την μετακίνησή μας εδώ είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να αλλάξουμε πλέον αυτό το συνήθιο να σταματήσουμε αυτή τη μόνιμη δαπάνη, να συνεδριάζουμε μόνο στις Βρυξέλλες, να εξοικονομήσουμε το, δι... και το δημόσιο χρήμα για καλύτερους στόχους. Ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος Ήτον χάρισε ένα λεπτό. Κάθε φορά ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο στο Στρασβούργο από ό,τι θα έπρεπε. Ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο στο Στρασβούργο. Είναι απαράδεκτο, κανένας δεν το κατανοεί αυτό. Δεν θα έπρεπε να επιλέγουμε να ερχόμαστε καθόλου στο Στρασβούργο. Θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα, ένα επιπλέον δικαίωμα, να αποφασίζουμε, εν πάση περιπτώσει, να επιλέξουμε που συνεδριάζουμε. Ο συνάδελφος κύριος Πόσολτ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα για τους πολιτικούς που ζουν κοντά στο Στρασβούργο, αλλά δεν είναι εύκολο να ερχόμαστε όλοι εδώ. Χρειάζεται μια μέρα για να έρθουν εκπρόσωποι από την εκλογική μας περιφέρεια. Υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε με το Στρασβούργο, ας το ξεφορτωθούμε έκθεση Μαγκίνες έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Χάναν. για την έκθεση Μαγκίνες για την Επιτροπή Αναφορών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα θέμα θα ήθελα να θέσω το σκάνδαλο των κατασχέσεων ε, γεών στην Ισπανία και ιδιοκτησιών στην Ισπανία. Ανεξαρτήτως της εθνικότητας ε, της εκλογικής μας περιφέρειας και της καταγωγής μας πάρα πολύ, υποφέρουν από τους νόμους αυτούς στις ισπανικές ακτές όπως και οι πολλοί χιλιάδες Ισπανοί ε, πραγματικά οι προσπάθειες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ εμποδίστηκε με απαράδεκτο τρόπο από τους Ισπανούς συναδέλφους. Και θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, συναδέλφους του Παρτίτο Ποπουλάρ να θυμούνται ότι είναι η ιδιοκτησία κάτι το οποίο θεωρείται ιερό και όσιο και δεν θα πρέπει τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία να φύγονται από οποιαδήποτε κρατική μη ρύθμιση. για την έκθεση Ζαμπόρσκα και την εισαγωγή της έννοιας του ε, φίλου. Ο κύριος Τάκουλα έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Τάκουλα είπα έχει ζητήσει το λόγο. Κοιτάξτε, όσον αφορά την έκθεση Ζαμπόρσκα, θα ήθελα να πω το εξή. Ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό η ισότητα των ευκαιριών να ισχύει και στο Κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη στι ε, επιτροπέ. Και όταν θα υπάρξουν οι καινούργιοι κατάλογοι σε σχέση με τι εκλογέ, είναι σημαντικό τόσο άντρε όσο και γυναίκε να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Είναι λοιπόν σημαντικό κάποια στιγμή να επιτύχουμε το στόχος μας όπου ε, το φύλλο να μην παίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο η τεχνογνωσία. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό στις ομάδες, τον να υπάρχουν πραγματικά ικανά άτομα και νομίζω ότι μόνο έτσι, μέσα από την τεχνογνωσία, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Έκθεση Μόργαν, κοινοί κανόνε για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπορούμε να κάνουμε σημαντική εξοικονόμηση αν συστήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλέγμα, ένα δίκτυο. Ε, κάποια στιγμή, ε, όπου πολλές στιγμές στην Ευρώπη υπάρχει πλεόνασμα ενεργειακό και εάν λοιπόν ε, μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό δίκτυο, αυτό θα περιορίσει και την κατανάλωση ενέργειας. Δυστυχώς η ελεύθερη αγορά ε, Δυστυχώς δεν την υπερψηφίσαμε σε αρκετές εκθέσεις σήμερα. Εμείς ακολουθούμε την εναρμόνιση, τις σταθερές τιμές, την ε, διαπραγμάτευση των θέσεών μας απέναντι στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες. Όμως εδώ υπάρχει μια σημαντική ιδεολογική διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα σε μια ελεύθερη αγορά που θα βασίζεται στην αμοιβαιότητα και σε μια εναρμονισμένη αγορά που θα αφορά στην επιλογή των καταναλωτών. Θεωρώ λοιπόν ότι ελοχεύουν σημαντική κινδύνη για μια χώρα όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία. Εμείς ήμασταν ε, ε, καθαροί παραγωγή μέχρι πριν από δύο χρόνια και τώρα ε, και εμείς ε, δυστυχώς δεν είμαστε ε, πλέον εποφελούμενοι. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία είναι καθαρός σε συνεισφορές και δεν αποκομίζει το ωφέλη που θα έπρεπε. Κύριος Καμάλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν προχωρήσω θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στην εισηγήτρια την κυρία Μόργαν η οποία δεν θα είναι πλέον υποψήφια ε, νομίζω θα συμφωνώ όλοι ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με αυτή την έκθεση. Αν δούμε λιγάκι την ιστορία της απελευθέρωσης στις τηλεπικοινωνίες, έχουμε ένα μεγάλο επίτευγμα όσον αφορά την επιλογή, της ε, τιμές, ε, τις καλύτερες υπηρεσίε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ντροπή το ότι για τα ταχυδρομεία και την ενέργεια δεν επιτέχθηκε το ίδιο. Ε, σαφώς ε, γίναν κάποια σωστά βήματα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της ε, αποσύνδεσης και των δικτύων. Δεν είναι σωστό ορισμένες αγορές όπως αυτή της Μεγάλη βρετανία, να είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό ενώ η ε, Γερμανία και η Γαλλία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμά, όμω εμποδίζουν το να μπούμε εμεί στι δικέ του αγορέ. Πλέον έχει περάσει η εποχή του προστατευτισμού και έχει φτάσει η στιγμή να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά. Πάμε στην ε, επόμενη έκθεση, στην Μπελέτ. Για τα ελαστικά, ε, για τα ελαστικά, εν πάση περιπτώσει, έχει το λόγο ο κύριος Τάκουλα εκ νέου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ε, ότι θέλω να αποτύσω ένα φόρο τιμή στην έκθεση του Ιβο Μπελέτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, χρειάζεται εξοικονόμηση ενέργεια στι μεταφορέ και ταυτόχρονα να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο αποτελεσματική. Είναι σημαντικό λοιπόν να μιλάμε για τα επίσωτρα, τα ελαστικά. Ε, όταν όμως μιλάμε για οδικές μεταφορές και ελάστιχα στην έκθεση θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι τίθεται ένα θέμα ασφαλείας. Η οδική ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ισορροπία. Όταν κάνουμε τέτοια ε, ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να γίνονται με το σωστό τρόπο, με εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά αυτό να μην είναι ει βάρο τη οδική ασφάλειας. Δεν μπορεί να θυσιαστεί ε, και ούτε σπιθαμή να δώσουμε σε αυτή την υπόθεση της οδικής ασφάλειας. Ε, γνωρίζουμε ότι είναι η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή. Relazione Valean. Modifica regolamento 717 sulla Έκθεση Βαλεάν, τροποποίηση κανονισμού για την ε, κινητή τηλεφωνία και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και πάλι κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Βαλεάν. Πάρα πολύ καλή η έκθεσή της, οφείλω να σας πω. Και είναι επίσης ζωτικής σημασία στην Ευρώπη, στο μέλλον, να έχουμε μια εσωτερική αγορά όπου παντού όμως στην Ευρώπη να υπάρχει δυνατότητα μείωσης ε, των διεθνών κλίσεων, των τιμών. Ε, όλοι ταξιδεύουμε από χώρα σε χώρα και βλέπουμε ότι χρειάζεται να αγοράσουμε άλλη κάρτα SIM ή να κάνουμε διάφορες ε, κινήσεις και ενέργειες για να χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο και τελικά πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας ε, ταξίδια. Αυτό περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει παντού να είναι ενιαία η κατάσταση και οι διεθνείς κλήσεις να μην κοστίζουν τόσο ακριβά για να είναι αντίστοιχη η χρέωση παντού. Θα πρέπει εδώ να προέχει το συμφέρον των πολιτών. Μόνο έτσι θα πετύχουμε μείωση των τιμών των διεθνών κλίσεων. Ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ω εισηγητή ε, για τα θέματα τη ιστορική αγορά ε, είμαι πολύ υπερηφανό ε, για το ότι κατορθώσαμε να επιφέρουμε μεγάλη διαφάνεια. Ένα από τα προβλήματα τελευταία χρόνια ήταν ότι οι καταναλωστές όταν γυρίζουν σπίτι του διαπιστώνουν ότι έχουν πληρώσει παραπάνω χρήματα από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχει το θέμα λοιπόν τη διαφορά των τιμών και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν υπήρχε αυτό ο κανονισμό θα έπεφταν οι τιμέ έτσι κι αλλιώ. Η Κομισιόν έχει ομολογήσει ότι οι περισσότεροι ε, καταναλωτές ε, δεν χρησιμοποιούν την περιαγωγή. Εκείνο λοιπόν που κάνουμε είναι ότι ε, περιορίζουμε το κόστος για κάποιους επίλεκτους, για ευρωβουλευτές, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι εταιρείε όταν προσπαθούν να ανακτήσουν το κέρδος τους δεν θα καταφέρουν και θα εκμεταλλεύονται τους πολίτες. Δεν πρέπει να ληστεύουμε τους φτωχούς για να δίνουμε περισσότερα προνόμια στους πλούσιους. Ο κύριος Γκόλνης. Κύριε Πρόεδρε, εγώ χαίρομαι για την έκθεση της κυρίας Βαλεάν για ένα θέμα που ε, για αλλαγή οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται απολύτως σε αυτό το τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οφείλω να πω ότι η κατάσταση καμιά φορά είναι τελείως απαράδεκτη εξαπάτηση των καταναλωτών που εν εκπληκτοί διαπιστώνουν ότι αν έχουν χρησιμοποιήσει ένα κινητό τηλέφωνο σαν αυτό που λέει στη συνδρομή τους ότι ε, συμπεριλαμβάνεται και η διεθνής κίνηση και οι διεθνείς κλήσεις. Για παράδειγμα, σε ό,τι με αφορά πρόσφατα πήγα στην Ιταλία. Σε μια, μια μέρα μπήκα στο ίντερνετ με το τηλέφωνο μου δύο-τρεις φορές και ήρθε ο λογαριασμός της γαλλικής εταιρείας Orange που είναι ε, περίπου κρατική 1.200 ε, ευρώ. Μετά πήγα ε, στην Εβιάν και στη Γενέβη 3.000 ευρώ, πάλι σε μια μέρα. Μα είναι χαρακτήριστες αυτές οι ενέργειες. Είναι σκέτη απάτη και φταίνε αυτέ οι εταιρείε, δεν υπάρχει καμία διαφάνεια ε, ε, από την πλευρά των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να ενοποιηθούν οι κανόνε για τη διαφάνεια των συμβάσεων για να γνωρίζει ο κόσμο τι γίνεται με την κινητή τηλεφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς και είμαστε όλοι υπέρ των χαμηλότερου κόστους των κινητών. Κανένας δεν θα μπορούσε να είναι κατά. Αλλά αυτό είναι το ένα τμήμα της εξίσωσης. Όταν υποχρεώνουμε εμείς τις εταιρείες να χαμηλώσουν το κόστος, βρίσκουν τα χρήματα από αλλού και γι' αυτό αυξάνουν το κόστος των συνδιαλέξεων αυτών που δεν ταξιδεύουν. Δηλαδή, οι μη ταξιδεύοντες ε, βοηθούν τους ταξιδεύοντες. <clears throat> Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που έχουν να πληρώσουν περισσότερα τώρα για τα τηλέφωνά τους για να μπορούν οι ευρωβουλευτές, οι επίτροποι και γενικά οι πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες να ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο. Εμείς δεν είμαστε υπεράνω, όλοι έχουμε συμφέροντα από τη μείωση των συμφάσεων και των ρυθμίσεων που προωθούμε στον τομέα αυτό εδώ και ένα χρόνο. Για να καταλάβετε πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην Ευρώπη, διαβάστε <coughs> την έκθεση αυτή. Ποιος έχει την εξουσία και σε ποιον επιβάλλουμε την εξουσία αυτή. Εμείς οι Ευρωκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σφάιντερ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Ε, θέλω να σας πω ότι εγώ υπερψήφισα αυτήν την έκθεση γιατί πιστεύω ότι αυτά τα οποία έλαβαν χώρα στον τομέα της ε, ακίνητης περιουσίας είναι πολύ σημαντικά. Όταν άρχισα να δουλεύω στις ε, Βρυξέλλες ε, το ένα λεπτό κόστιζε 3 ευρώ και παραπάνω και τώρα λόγω αυτής της ρύθμισης πληρώνουμε πολύ λιγότερα ε, αυτό λοιπόν είναι ε, προς όφελος όλων των εταιριών στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι ε, το τιμολόγιο πολλές φορές ήταν ασαφές, τουλάχιστον κατά παρελθόν, κυρίως όσον αφορά τα μηνύματα, τα SMS. Τώρα, όσον αφορά την, τα τηλεφωνήματα, μειώθηκαν βέβαια οι τιμές. Μέχρι τώρα τα μηνύματα κόστιζαν πάρα πολύ. Και με αυτή τη ρύθμιση κάναμε ένα πολύ ε, σημαντικό καλό βήμα προς όφελος του ε, καταναλωτή. Σήμερα λοιπόν που είναι σημαντική η μεταφορά των ε, δεδομένων μέσα από τα κινητά θεωρώ ότι αυτά που πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι πολύ σημαντικά. Έκθεση ασφάλειας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σκίνερ. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Είναι τεράστια η προσπάθεια που πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό, αλλά νομίζω ότι η νομοθετική πρόταση είναι πολύ καλή. Είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί η Ευρώπη να συνεργαστεί και να βρει λύσεις στην κατανομή του βάρους και στην κάλυψη των αναγκών που βασίζεται στην οικονομική συνεργασία. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ποτέ να μην βιώσουμε μια τραπεζική κρίση όπως αυτήν την οποία βιώνουμε τώρα. Αυτό θα βοηθήσει επίσης και αυτούς οι οποίοι έχουν δυσκολίες στη δική μου χώρα να αποπληρώσουν τα στεγαστικά δάνεια για δύο χρόνια θα επιδοτηθούν. Θα πρέπει να δούμε πώς το πρόγραμμα αυτό θα προχωρήσει και αντίστοιχα να προσπαθήσουμε να ελαφρύνουμε τα βάρη τα οποία φέρει κάθε χώρα. Νομίζω ότι οι ίδιοι οι πιστοτικοί οργανισμοί στις χώρες μέλη να πάρουν μέτρα για να διευκολύνουν τους ε, ε, δανειοδοτημένους πελάτες τους όταν έχουν δυσκολίες στην επιστροφή του χρέους τους. Ευχαριστώ. Έκθεση Höckmark. Πυρηνική ασφάλεια. Δίνω το λόγο στον Ήτον Χάρις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Καμάλ που έκανε την εκατοστή παρέμβασή του στην Ολομέλεια από τότε που ήρθε εδώ. Κάποιοι από εμά εκπλήσονται γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να μιλήσει εκατό φορές ο κύριος Καμάλ. Συγχαρητήρια όμως για μια ακόμη φορά. Καταρχάς δεν μπορεί κανείς να είναι κατά της πυρηνικής ασφάλειας και όταν μιλάμε για την πυρηνική ασφάλεια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την ενέργειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το μέλλον. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει περισσότερη πυρηνική ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, στο ε, μέλλον. Έχω αρχίσει να συχαίνομαι πια αυτές τις ανεμογεννήτριες οι οποίες βιάζουν το περιβάλλον και δεν προσθέτουν τίποτα ε, στα εθνικά δίκτυα, δημιουργούν προβλήματα, δεν παράγουν ανανεούμενη ενέργεια αλλά κάποια επιπλέον ποσά ενέργειας όταν δεν χρειάζονται. Έκθεση Ρωμέβα για τον κοινοτικό έλεγχο ε, στον τομέα της αλίας. Ο Άλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει σαν στόχο τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλίας και να ελέγχουν γραφειοκρατικά τη χορήγηση αδειών ερασιτεχνικής αλίας κτλ. Είναι κάτι το οποίο πολύ σωστά προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις όχι μόνο από αυτούς που εμπλέκονται στον συγκεκριμένο τομέα αλλά από όλους όσους ενδιαφέρονται με την αλία και την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Και βλέπω ότι έγινε δεκτή η τροπολογία 48 ευτυχώς η οποία εν μέρη τουλάχιστον αποκαθιστά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών που αποφασίζουν για το αν θα πάρουν κάποια πρώτα βήματα για την αδειοδότηση της ερασιτεχνικής αλίας. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα είναι υπεύθυνα για να κρίνουν εφόσον υπάρχουν επιπτώσεις και στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν επιπτώσεις από τέτοιου είδους αλλιευτικές δραστηριότητες στα αλλιεύματα στο σύνολό τους. Την πάτησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της αυτή και η κακή πρόταση ε, εν ολίγης τουλάχιστον έχει βελτιωθεί θα έλεγα. Κύριος Χάναν, μετά από 10 χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο τίποτα δεν θα με εξέπλητε αλλά εγώ πραγματικά έχω εκπλαγεί από την πρόταση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής στους ερασιτέχνες αλλιείς οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν κάθε ε, αλλιεύμα σε σχέση ε, με το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις εθνικές ποσοστώσεις. Υπήρξε ένα σκληρός πόλεμος φθοράς από τους ε, Σκοτσέζους, τους Πατριώτες και τους Βρετανούς οι οποίοι ε, εκπροσωπούν τις περιοχές αυτές, τον κύριο Χάτσον, τον κύριο Στίβενσον και άλλους και τον Άλιστερα από τη Βόρεια Ιρλανδία ο οποίος θέλει να γίνουν σεβαστές οι παραδόσεις των κοινοτήτων μας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εφαρμόζουμε τους υπάρχοντες κανονισμούς. Και η μοναδική μας προσπάθεια εδώ είναι όχι να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας σε νομικό επίπεδο, αλλά να ομοθετήσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν είναι σωστό όμω το να ψηφίσουμε νέου νόμου. Θα πρέπει να εξαντλήσουμε τι νομικέ δυνατότητε, τι οποίε έχουμε στη διάθεσή μα πρώτα. Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με την έκθεση αυτή περί ανανοήσιμων πηγών ενέργειας θέλω να πιστεύω ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες, οι τροπολογίες ε, ε, πέρασαν, κάποιε άλλε απορρίφθηκαν. Η τροπολογία 49 πέρασε με 500 τόσους ψήφους, με 54 μόνο κατά και η 50 υποστηρίχθηκε. Η 2 πέρασε, ήταν βέβαια σε μπλοκ με την 11 και την 7 και η 92 κατέπεσε, η 93 επίση κατέπεσε ε, και αυτό κατ' ουσίαν ζητάμε. Το επόμενο βήμα είναι τι θα κάνει τελικά το Συμβούλιο με το άρθρο 47. Ε, μήπως ε, θα έχει ε, διαφορετική προσέγγιση. Σήμερα δεν είναι κανείς εδώ από το Συμβούλιο για να απαντήσει. Όμως η μεταρρυθμίση δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αλλάξουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική. Και θέλω να πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα αδράξουν ευκαιρία για να στείλουν την πράσινη βίβλο σε όσο δυνατόν περισσότερες εκλογικές περιφέρειες για να εισακουστεί η φωνή τους. Έκθεση Βίσερ, διατήρηση των αλληλευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων. Ο κύριος ε, Καμάλ που τώρα πια θα κάνει την εκατοστή πρώτη παρέμβασή του, αφού την έκανε την εκατοστή. Ε, είναι λοιπόν ε, πράγματι ορόσημο το να φτάνω στην εκατοστή πρώτη παρέμβασή μου. Ε, αυτή η έκθεση έχει ενδιαφέροντα τίτλο. Ε, αναφέρεται στη διατήρηση των λεπτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων. Και θέλω να πω ότι αν πραγματικά θέλουμε τα βέλτιστα τεχνικά μέτρα για να διατηρούμε του αλευτικού πόρου, αυτά δεν υπάρχουν στην κοινή αλευτική πολιτική υπάρχουν τα αποτελέσματα της κοινή ελευτικής πολιτικής που δείχνουν ότι είναι αποτυχία όσον αφορά τους ελευτικούς πόρους. Ε, έχει πια οριμά στιγμή για να αναθεωρήσουμε ε, την κατάσταση. Ας δούμε τι γίνεται με την Ισλανδία. Εκεί έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα που μπορούν να μεταφερθούν ή στη Νέα Ζηλανδία τα δικαιώματα αλληλείας ε, κληρονομούνται από γενιά σε γενιά. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι αν εμπιστεύεται κανείς στην αγορά κράτος δικαίου, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Αυτό πολύ συχνά είναι πολύ καλύτερη λύση από αυτό το σοβιετικό, σοβιετικό μοντέλο της κοινή ελευτικής πολιτικής που αποδείχθηκε ότι είναι μια καθαρή αποτυχία. Ευχαριστώ έκθεση Μπούσουτιλ για την κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη. Έχει το λόγο ο ίδιος ο εισηγητής. Όχι. Κάποια κυρία φωνασκή αλλά χωρίς μικρόφωνο. σας έστειλα ένα μήνυμα γραπτό για την έκθεση Φίσερ. Ήθελα κάτι να πω και για την έκθεση Φίσερ, αλλά πήρατε μήνυμα. Δεν πήρατε μήνυμα για την έκθεση Φίσερ. Όχι. Δεν πήρα τίποτα. Όχι, δεν πήρα τίποτα κυρία Βάιντερ, προβλέπεται η εγγραφή για τις ε, επεξηγήσεις ψήφου να έλθουν στο Προεδρείο πριν ξεκινήσουν οι επεξηγήσεις ψήφου. Εγώ σας έδωσα το λόγο στην προηγούμενη έκθεση, αν και δεν είχατε λάβει το λόγο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω δεύτερη φορά, γιατί θα βλάψω τους συναδέλφους οι οποίοι περιμένουν να πάρουν το λόγο. Λοιπόν, δεν ήλθε κανένα αίτημα για επεξήγηση ψήφου από πλευρά σα. Ευχαριστώ, κύριο Μπούσουτιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για να εξηγήσω πώς ψήφισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην έκθεσή μου. Για την κοινή μεταναστευτική πολιτική υπήρχε η έκθεση αυτή καθ' αυτή και ένα εναλλακτικό ψήφισμα. Ψηφίσαμε να βγει μια παράγραφος που είχε μπει από το σοσιαλιστικό μπλοκ στην έκθεσή μας. Για να δώσουμε δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες. Εμείς δεν συμφωνούμε με τέτοια μέτρα. Γι' αυτό ψηφίσαμε διαφορετικά στην Επιτροπή και δυστυχώς ε, ε, και ε, δεν πέρασε ούτε στην Ολομέλεια. Θα μπορούσε να έχει βγει αυτή η παράγραφος από την έκθεσή μου. Εν πάση περιπτώσει, Τελικά υπερψηφίσαμε την έκθεση γιατί θεωρούμε ότι είναι καλή και περιλαμβάνει καλό πρόγραμμα και τις θέση του Κοινοβουλίου για την κοινή μεταναστευτική πολιτική. Κύριος Γκολνής. Ευχαριστώ. αρχή, δράση, εργαλείο για μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Τεράστιο χώρο καλύπτει και πεδίο εκθέση Μπουσούτιλ. Οι αρχή, αρχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει χρειάζεται επιπλέον 60 εκατομμύρια εξοκοινοτικούς μετανάστες μέχρι το 2050. Μα παρά ε, τα εκατομμύρια ανέργων που έχουμε και φτωχών, μαζικές απολύσεις, κλείσιμο εταιριών οι δράσει ποιε είναι όλο και περισσότερα δικαιώματα να έχουν οι μετανάστε και οι πληθυσμοί του, ιδιαίτερα το δικαίωμα ψήφου και απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά εργασία και στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Τα εργαλεία ε, θετική διάκριση, αναγνώριση άτυπων προσόντων, όποια και να είναι αυτά, ενώ από του Ευρωπαίου απαιτούμε διπλώματα και τίτλου, αναγωνισμένους. Νέα κατηγορία, λέει, περιβαλλοντική μετανάστε και αναγνώρισή τους και υποχρέωση για του ευρωπαϊκού λαού να ε, ε, προσαρμοστούν στην αναπόφευκτη ε, πλημμύρα που οργανώνουμε και εμείς μεταναστών. Θα πρέπει τα μεσανευτικά ρεύματα να οργανηθούν, να ε, έχουμε και πάλι τα εσωτερικά σύνορα, οικογενειακή πολιτική για ανανέωση, δημογραφική, ευρωπαϊκή, να επιβληθεί η εθνική και ευρωπαϊκή προτίμηση παντού. Ο κύριος Μποργέζιο. Ε, Έχω πολλές επιφυλάξεις για την έκθεση αυτή. Όπως είπε και ο προηγούμενος, η πρόβλεψη αυτή είναι πολύ απογοητευτική. Τη στιγμή που έχουμε προβλήματα ανεργίας για εκατομμύρια εργαζομένους και έχουμε, προβλέπουμε 60 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια είναι πραγματικά εξωπραγματική η πρόβλεψη αυτή. Τη στιγμή που εμείς συζητάμε για το πώς θα ρυθμίσουμε πώς θα οργανώσουμε το μέλλον της μετανάστευσης συμβαίνουν ε, ε τραγωδίες. Κάποιες από αυτές ε, βοήθησε η χώρα μου να ξεπεραστούν βέβαια, να αποφευθούν, όπως ε, το τουρκικό σκάφος, εμπορικό σκάφος Πιλάρ με τους μετανάστες που σώθηκαν από Ιταλική παρέμβαση. Η Μάλτα δεν έχει παίξει το ρόλο που έπρεπε δεν έχει υποδεχθεί όπως θα έπρεπε ε, τους μετανάστες αυτούς και δεν έχει αντιμετωπίσει ε, τα σκάφη που προέρχονται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Εμείς δεν τα καταφέρνουμε με το κέντρο υποδοχής της Λαμπεντούσα, το οποίο όπως όλοι γνωρίζετε πλέον έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες υποδοχής τις οποίες έχει πρέπει η Ευρώπη να παρέμβει, να καθορίσει τους συγκεκριμένους κανόνες. Ζητάμε μια ουσιαστική αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τη δική μου χώρα για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Ας ξυπνήσει η Ευρώπη. Φυσικά πρέπει να υπάρξουν κανόνες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ρεύματος. Τελευταία επεξήγηση ψήφου, αν και δεν είχε έρθει επίσημα το αίτημα εγκαίρως, η κυρία Βάιμπερ να μας εξηγήσει για ποια έκθεση θέλει να κάνει τη δήλωσή της. Σας είπα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, ε, ότι ήθελα να κάνω μια επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Βίσερ της Επιτροπής Αλίας. Πρόκειται για τις δυνατότητες Ε, τις αλλιευτικές. Η χώρα μου, Πρόεδρε, ξέρετε, η Λετωνία, έχει 550 ε, χιλιόμετρα ακτές Έχουμε 8 ευρωβουλευτέ και δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε όλε τι επιτροπέ, Γι' αυτό ε, η αλία όμω είναι πολύ σημαντική για τη Λετωνία και για την παραδοσιακή μα οικονομία. Η έκθεση δεν ασχολείται ε, επαρκώ με την προστασία τη παράκτεια αλίας. Ξέρω ότι είναι τεράστια τα προβλήματα, αλλά η υπερβολική ρύθμιση τελικά πού οδηγεί. Απειλείται η παράκτεια παραδοσιακή αλία και κινδυνεύουν οι αλληλείς τη Βαλτική να εκδιωχθούν από τη θάλασσά τους. Ε, οφείλει λοιπόν το Κοινοβούλιο να φροντίσει οι χώρες που βρέχονται από τη Βαλτική να σεβαστούν και τις παραδοσιακές μεθόδους αλίας και την παραδοσιακή ε, οικονομία και αλία. Διότι τώρα έρχονται αλίες μεγάλες εταιρείες και αγοράζουν τα χώρια που έχουμε και χάνουν τη δουλειά του οι άνθρωποι και τα ψάρια έρχονται από τον ωκεανό. Ολοκληρώσαμε εδώ τις επεξηγήσεις ψήφου. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Σα ευχαριστώ πολύ.